So, meine sehr verehrten και κύριοι, είμαστε σε μια κάπως δύσκολη κατάσταση. Έχουμε περάσει το ακαδημαϊκό τέταρτο, το χρόνο αναμονή των επιβλημένο και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο για την ημερήσια διάταξη. Αλλιώς θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε. Αλλά δεν έχω απαρτία. Και έτσι προτείνω να ξεκινήσει η παρουσίαση όσοι ενδιαφέρονται, φαντάζομαι είναι ήδη εδώ. Να, την παρακολουθήσουμε λοιπόν και αναλόγως θα πράξουμε για τα υπόλοιπα και τις αποφάσεις που έχουμε λάβουμε στη συνέχεια. Και έχω το εξής πρόβλημα με την, με την ημερήσια διάταξη. Ε, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τα σημεία 1, 2, 3, 4 αφού δεν έχουμε απαρτία ένα, δύο, τρία μάλλον και προτείνω να δούμε την παρουσίαση μελέτη σχετικά με την απενεργοποίηση της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τους εκπροσώπους του Policy Department. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ο κύριος Τζουζέ Πεντεπάλο, καθηγητής Τζουζέ Πεντεπάλο από τη Yams International. Ευρωπαίος ειδικό στα θέματα της διαμεσολάβησης, ο οποίος έχει εκπονήσει και τη μελέτη για τη διαμεσολάβηση. Θα έλεγα λοιπόν να του δώσουμε κατευθείαν το λόγο. Καθηγητή Δεπάλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Καλησπέρα σε όλου. Έχω ξανάρθει για να μιλήσω για διαμεσολάβηση. Άρα, είτε αυτά που είπα κατά το παρελθόν ήταν αρκετά σαφή, είτε αυτά που είπα είναι και τόσο άσχημα. Για οποιοδήποτε λόγο με ξανακαλέσατε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Όπως θα βλέπετε από τον τίτλο της μελέτης που μου ανετέθη από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων το περσινό καλοκαίρι, η οδηγία για αυτή τη διαμεσολάβηση χρειάζεται εκείνης από την αρχή, σαν ε, τον υπολογιστή. Διότι όπως γνωρίζετε και ξέρει η Επιτροπή, ο αντίκτυπος εφαρμογής της στα κράτη-μέλη υπολείπεται των προσδοκιών. Αναφέρομαι σε προφορική ερώτηση που εσείς κύριε Πρόεδρε υποβάλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί στην Αντιπρόεδρο την κυρία Vivian Redding το Δεκέμβριο του 2012. Μας ρωτήσατε τι ρωτήθηκε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του το περιορισμένου ρυθμού των περιπτώσεων διαμεσολαβήσεων στα πλαίσια του αστικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλαξα τη διαφάνεια στην οθόνη, συγγνώμη, άλλαξα τη σειρά των διαφανειών που βλέπετε στην οθόνη. Παρουσιάζω τη μελέτη και τη δομή της. Μα ζήτησε το Κοινοβούλιο να του πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τον αριθμό 2. Δηλαδή να κάνουμε μια ανάλυση της νομοθεσίας που εφαρμόζει την οδηγία για τη μεσολάβηση στα κάτι μελη και εμείς ε, προτείναμε στο Κοινοβούλιο να εξετάσουμε τα κάτι μελη η δεύτερη ερώτηση, υπαριθμόν 3. Μα ζήτησε το Κοινοβούλιο βάσει τη έρευνα των θετικών αποτελεσμάτων, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά όσον αφορά την εθνική νομοθεσία. Με βάση αυτό, αν θα μπορούσαμε να προτείνουμε νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, ούτω ώστε να πετύχουμε το σκοπό, δηλαδή την εφαρμογή. Τρίτον σημείο, το υπαριθμόν ένα εδώ στη διαφάνεια, κάτι που αποφασίσαμε να κάνουμε οι ίδιοι. Ρωτούσαμε τον κόσμο στην Ευρώπη τι γίνεται να σχολιάσει την ομοθεσία του. Άρα θεωρήσαμε ότι έπρεπε να επικαιροποιήσουμε την έρευνα για το κόστος της έλλειψης διαμεσολάβησης. Τι θέλαμε να κάνουμε. Το παράδοξο της διαμεσολάβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει η κασία ότι είναι πολύ αποτελεσματική διαδικασία που τη χρησιμοποιούν ελάχιστοι. Και αυτό είναι το παράδοξο, γιατί είναι πολύ αποτελεσματική, πολύ καλή, αλλά ελάχιστοι τη χρησιμοποιούν. Λοιπόν, το 2011 είχα την τύχη να παρουσιάσω εδώ την έρευνα. Στόχος της να παριθμίσει και να αποστοτικοποιήσει αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή ότι μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο και χρήματα με τη μεσολάβηση. Το θέμα ήταν πόσο. Ποιο είναι το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση και να μην χρησιμοποιείται αρκετά. Τα αποτελέσματα της μελέτης τα έχουμε επικαιροποίησει. Δεν θα σας δείξω παλιά στοιχεία, αλλά εν συντομία τα νέα. Είναι εκπληκτικά τα αποτελέσματα, διότι τι βλέπουμε. Αν χρησιμοποιεί το διαμεσολάβηση, ας υποθέσουμε συνεχώς μέσω ρυθμιστικής παρέμβασης, σε κάθε περίπτωση, πριν υπάρξει προσφυγή στα δικαστήρια του αστικό δίκαιο. Θα αρκούσε 19% των διαμεσολαβήσεων να εφαρμοστούν. 19 επιτυχείς, 81 να αποτύχουν, δηλαδή να εκδικάζονται. Εάν 19 ε, πετύχαναν, θα γλιτώναμε χρόνο. Κόστος. Αν οι επιτυχείς διαμεσολαβήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε υπόθεση αστικού δικαίου, ήταν 24%, θα γλιτώναμε κόστος και είναι το σημείο ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Δηλαδή, ποιο είναι ο ελάχιστο αριθμό διαμεσολαβήσεων που θα πρέπει να λάβει η χώρα, ώστε τα ωφέλη που απορρέουν από την επιτυχή διαμεσολάβηση και δεν υπάρχει δίκη, εξισορροπούνται από τι απώλειε των διαμεσολαβήσεων που δεν πάνε καλά. Δηλαδή, ο κόσμο προσφεύγει στη διαμεσολάβηση, δεν λειτουργεί και πάει στο δικαστήριο. Γιατί οι επιδόσεις μεσολάβησης είναι τόσο υψηλές. Διότι η μικρή αύξηση του κόστους, είναι πολύ μικρή η αύξηση του κόστους για τις αποτυχημένες διαμεσολάβησεις, κυρίως όταν είναι δωρεάν διαμεσολάβηση. Είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα των κερδών, των ωφελών κάθε επιτυχίας, κάθε επιτυχούς διαμεσολάβησης. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια διαδικασία που πράγματι μπορεί να έχει ύψιστες επιδόσεις ακόμα και αν το ποσοστό των επιτυχιών είναι τόσο χαμηλό όπως προανέφερα. Όπως σας είπα, αποφασίσαμε ότι το πρώτο βήμα που θα κάνουμε πριν αναλύσουμε την νομοθεσία θα ήταν να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Χάρη στη βοήθεια της Diana Wallis και άλλων πυρογνωμόνων παρόντων, Ετοιμάσαμε ένα αρκετά αναλυτικό ερωτηματολόγιο, 45 ερωτήσεις και ζητήσαμε από τους εμπειρογνώμονες να μας δώσουν μια εικόνα για τη χώρα τους. Βλέπετε, είναι αρκετά μικρό το διάγραμμα, λάβαμε απαντήσεις από όλα τα κράτη-μέλη, περίπου 30 κατά χώρα, ε, με σημαντικά ακραία σημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα και στη Ρουμανία. 210 απαντήσεις αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διαμεσολάβησης στις χώρες. Όλες οι χώρες εκπροσωπηθήκαν 816 απαντήσεις, πολύ μεγάλος αριθμός απαντήσεων. Όταν ζήτησε απάντηση για πράσινη βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια χρόνια για την οδηγία, περίπου 150 ερωτήσεις κατέφτασαν. Άρα η αύξηση απαντήσεων δείχνει ότι η οδηγία πρόθεσε την όλη συζήτηση για τη μοσολάβηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όσον αφορά το σημαντικό ερώτημα, το παράδοξο, ζητήσαμε του εμπειρογνώμονες να μας πούν ποιο είναι ο εκτιμόμενος αριθμός αναέτος των διαμεσολαβήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, τα σημαντικότερα στοιχεία δεν είναι στο διάγραμμα και ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Ότι σε αρκετές χώρες πολλοί κόσμος δεν είχε ιδέα για πόσε δημοσιολαβήσει είχαν λάβει χώρα. Είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί πολιτική για ένα φαινόμενο που δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία. Αυτό που βλέπετε είναι εκτιμήσει αλλά να έχετε υπόψη ότι 30, 40, 50, 60 ε, ρωτήσαμε κάποιες φορές να μας δώσουν απαντήσεις και βγάλαμε μέσο όρο. Άρα είναι σχετικά τα στοιχεία που βλέπετε. Όπως βλέπετε υπάρχει σημαντικός αριθμός χωρών, 46% των χωρών, όπου υπάρχουν λιγότερες από 500 διαμεσολαβήσεις την ημέρα. Άρα η διαμεσολαβήση που είναι 0,01% αριθμός δημοσιολαβήσεων που χρησιμοποιείται εδώ ποσοστό σε σχέση με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις. Μόνο τέσσερις χώρες που βλέπετε πάνω, ο αριθμός των δημοσιολαβήσεων είναι πάνω από 10.000 το χρόνο, το χρόνο έχει την ημέρα. Ε, τι σημαίνει. Αν ξεχωρίσετε τα στοιχεία, δεν είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα, διότι η μόνη χώρα η οποία έχει πάνω από 200.000 δημοσιολαβήσεις που έχουν ξεκινήσει σε ένα χρόνο είναι η Ιταλία, ενώ οι άλλες τρεις χώρες, η Γερμανία, Νεωμένο Βασίλειο και Ολλανδία, έχουν λίγο παραπάνω από 10.000. Διότι κάποιοι, σε κάποιες χώρες είπαν ότι είχαν πάνω από 10.000 υποθέσεις το χρόνο, κάποιοι άλλοι στις ίδιες χώρες είπαν ότι υπάρχουν λιγότερες από 10.000 το χρόνο. Άρα μαντεύουμε ότι ο αριθμός στρέφεται, είναι περίπου 10.000. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που περιέγραψα, δηλαδή το κόστος μη διαμεσολάβησης, τι κάναμε μαζί με τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων. Διασταυρώσαμε δύο ομάδες στοιχείων. Πήραμε την έκθεση για τη δημοσίευση του, της Παγκόσμιας Τράπεζας όπου εκεί για 190 χώρες αναφέρει τη διάρκεια και το κόστος της διαφοράς. Της διαφοράς της. Πήραμε λοιπόν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δίπλα σε αυτά τα στοιχεία, διάρκεια, κόστος της εκδίκασης στο αστικό δικαστήριο. Βάσει των στοιχείων που μας έδωσαν οι εμπειρογνώμονες, ρωτήσαμε τους εμπειρογνώμονε πόσο χρόνο και πόσες μέρες θα χρειάζεται για να λυθεί η ίδια διαφορά. Αν η διαμεσολάβηση γίνει πριν την αποτυχία της εκδίκασης, έχουμε αύξηση σε κέρδος χρόνου και κόστος. Όταν επιτυχεί η διαμεσολάβηση, έχουμε κέρδος. Για να βρούμε στοιχείο αριθμητικό, Πρέπει να δούμε το ποσοστό τη διαμεσολάβηση. Ακολουθήσαμε μια πρώτη, ένα πρώτο σενάριο. Αν βασιστούμε στοιχεία τη Παγκόσμια Τράπεζα και έχουμε 566 ημέρε μέσω χρόνου διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθεια δείχνει διαφορά, αν όλε οι αστικέ υποθέσει πρώτα αντιμετωπιζόταν μέσω τη διαμεσολάβηση και η διαμεσολάβηση είχε επιτυχή αποτελέσματα σε μία περίπτωση από τις δύο, τότε η δίκη της οποίας προηγήθηκε ε, διαμεσολάβηση θα διαρκούσε 426 μέρες. Δηλαδή υπάρχει διαφορά με το... Θα γλιτώναμε 240 μέρες σε σχέση με την άλλη υπόθεση που εκδικάζεται χωρίς να έχει γίνει η διαμεσολάβηση. Τώρα, εάν 70% έχουν επιτυχείς διαμεσολαβήσεις και εφαρμόζονται πάντα διαμεσολαβήσεις, εκεί έχουμε μεγαλύτερες οικονομίες και έχουμε 212 ημέρες διάρκεια. Μετά είδαμε την, ε, την έκθεση της Επιτροπής ΕΠΑΖ του Συμβουλίου της Ευρώπης έκανε συντηρητική εκτίμηση και είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τον αστικό και τον εμπορικό έχουμε 13 εκατομμύρια υποθέσεις κάθε χρόνο, νέες υποθέσεις. Αν η οικονομία με ποσοστό επιτυχίας 50% είναι 240. Κάθε φορά που, που ε, ε, αναλύεται υπάρχει δημοσιολάβηση γλιτών 240 μέρες και βάζουμε αριθμό ε, υποθέσεων επί των ημερών που εξοικονομούμε, έχουμε γλιτώσει, έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια χρόνια ο χρόνος που πρέπει να περιμένουν οι διάδικοι για ένα χρόνο πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Λοιπόν, 8 εκατομμύρια χρόνια περίπου μπορούμε να γλιτώσουμε πλευρά χρόνου. Πολύ σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο. Μας δείχνει το μέσο κόστος της διαφοράς σε ευρώ με βάση την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. 9.179 είναι το μέσο κόστος της ε, διαφοράς. Εδώ αν υποθέσουμε ότι έχουμε 50% επιτυχία, ποσοστό επιτυχίας, το μέσο κόστος θα μειωθεί, θα πάει κοντά στο 8.000 και αν υποθέσουμε υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας της διαμεσολάβησης, το μέσο κόστος της διαφοράς θα μειωθεί ακόμα παραπάνω. Βλέπετε εδώ τις οικονομίες, το ποσοστό επιτυχίας 50% και είναι αρκετά συντηρητική εκτίμηση. Το 50% είναι αρκετά ε, συντηρητική προσέγγιση βάσει των στοιχείων. Για κάθε διαφορά τις οποίες προηγείται δημοσιολάβηση, κατά πό... Ε, είτε επιτυγχάνει είτε αποτυγχάνει, γλιτώνουμε πάνω από 1.200 ευρώ ανά υπόθεση. Και αν κάνουμε τους υπολογισμούς όπως και πριν, καταλήγουμε σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε. Γιατί λέω ότι είναι συντηρητική εκτίμηση, διότι η έκθεση σε ΠΑΖ, σε ΠΕ μάλλον, από εκεί που αντλούμε εμείς το στοιχείο για 13 εκατομμύρια διαφορές, δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη διαφορών, 1,5 εκατομμύρια στικές υποθέσεις ε, κατατίθενται στο ειρηνοδικείο κάθε χρόνο και δεν λαμβάνονται υπόψη από την έκθεση σε ΠΕΣ. Γι' αυτό είναι συντηρητική προσέγγιση. Δηλαδή οι οικονομίες θα μπορούσαν να είναι ακόμα ε, μεγαλύτερες. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα που βασικά ακολουθήσαμε τον καπνό, ούτως υπήν, για να εντοπίσουμε πού βρίσκεται η φωτιά. Όπως λένε οι Αμερικάνοι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λοιπόν, προσπαθούσαμε να δούμε τον αριθμό των ε, διαμεσολαβήσεων και προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι η φωτιά. Δηλαδή, ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο που δημιουργεί αυτού του αριθμού, παρέχει του αριθμού. Λοιπόν, ποια ήταν η υπόθεση. Όταν προστατεύεται ο εμπιστευτικό χαρακτήρα, η εμπιστευτικότητα και κινούνται, είναι πιο δραστηριοποιημένοι οι δικαστέ και είναι εύκολο να εφαρμοστούν οι συμφωνίε διαμεσολάβηση ή υπάρχουν οικονομικά κίνητρα ή κάτι τέτοιο. Ή οι νομικοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν του πελάτε για τη μεσολάβηση και η ποιότητα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης ε, ε, είναι εγγυημένη λόγω πολλού καλού συστήματος ε, που ελέγχει το σύστημα, που όλο σύστημα. Άρα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αν είναι αδύνατες οι μεταβλητές αλλού θα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Θέλαμε να δούμε πώς λειτουργούν τα αποτελέσματα λόγω των παραγωμένων, βάσει των παραγωμένων υποθέσεων. Το συμπέρασμα ήταν καμία, κανένα από τα χαρακτηριστικά αυτά θα λειτουργούσε και σε χώρες που υπάρχει μεγάλη προστασία. Οι δικαστές είναι πολύ δραστήριοι και εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν υπάρχουν πολλές διαμεσολαβήσεις όπως είδατε πριν. Είδατε τον πίνακα που ανέφερε τον αριθμό των διαμεσολαβήσεων. Δηλαδή η απόδειξη ότι κανένα από τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα παράγει Τα στοιχεία αυτά που είδαμε είναι όταν ρωτήσαμε ένα από τα δεύτερα ερωτήματα ποιο είναι το αποτελεσματικότερο νομοθετικό μέτρο που θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των δημοσιολαβήσεων στη χώρα σας. Και όπως βλέπετε, τα ανώτερα τα ε, μέτρα, πρωτοβουλίες που θα αύξανε τον αριθμό, είναι υποχρεωτική δημοσιολάβηση και υποχρεωτική ενημέρωση για τι διαμεσολαβήσει. Πριν κανεί προσφύγει στο δικαστήριο και να μπορεί να φτάσει στο δικαστή, είτε θα πρέπει να δοκιμάσει τη διαμεσολάβηση πρώτον, ή δεύτερον θα πρέπει να καθίσει με κάποιο σύμβουλο και να μιλήσει μαζί του και να ζυγίσει κανεί τα υπέρ και τα κατά τη διαμεσολάβηση ή μη διαμεσολάβηση στη διαφορά. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία πιο προσεκτικά, βλέπουμε ότι το καλύτερο μέτρο όμω δεν είναι υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε κάποιε υποθέσει διότι ρωτήσαμε να μας πούν οι εμπειρογνώμονες όχι μόνο ποια είναι τα ωφέλη κάποιων μέτρων, αλλά ποια και τα αρνητικά στοιχεία. Και σε κάποιες χώρες η επιλογή 1, υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θεωρείται σαν κάτι θετικό. Βέβαια πήραμε το μέσο όρο. Και είδαμε δύο μέτρα, υποχρεωτική ενημέρωση και υποχρεωτική διαμεσολάβηση με δυνατότητα αυτοεξαίρεσης, opt-out. Να σας εξηγήσω τι είναι. Και αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε το μέτρο που κερδίζει. Τι έχουν σαν κοινό οι δύο επιλογές. Δεν ζητούν από τα διάδικα μέρη να προβούν σε πλήρη διαμεσολάβηση και να πληρώσουν. Ζητούν από τα δύο μέρη να, τα μέρη να καθίσουν, να μιλήσουν με ένα σύμβουλο και τον ίδιο το διαμεσολαβητή στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση τότε αυτοεξαίρεση για να μιλήσουν, να, να προσπαθήσουν να βρουν λύση. Αν τα μέρη δουν ότι έχει πιθανότητες να έχει αποτέλεσμα η μεσολάβηση, μπορούν να αποφασίσουν να συνεχίσουν και να πληρώσουν. Εάν δεν θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα μεσολάβηση, μπορούν να αποσυρθούν. Το σύστημα βασίζεται επί της αδράνειας. Δηλαδή, περνάει ο κόσμο στη διαδικασία διαμεσολάβηση χωρί να είναι υποχρεωμένοι να φτάσουν μέχρι τέλου εκτό αν το επιθυμούν. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό γιατί, όπως είπα, δίνει στα μέρη μια σχετική εμπειρία στη διαμεσολάβηση και έχουμε εδώ και μια ε, εθνική τάση της διαμεσολάβησης η οποία αναπτύσσεται τώρα θα σας ε, πω ότι το πρώτο ενστικτό των ανθρώπων αλλά και των ζώων δεν είναι να διαμεσολαβούν αλλά να επιθύθονται. Τώρα, τι γίνεται με τα μη νομοθετικά μέτρα, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει που θα είναι εκτός της νομοθεσίας. Θα σας δείξω τα κύρια που είναι στην κορυφή. Στην έκθεση περιλαμβάνεται το Ζητήσαμε του εμπειρογνώμονε ε, βάσει τη αποτελεσματικότητα να ταξινομήσουν από τα πολύ αρνητικά στα πολύ θετικό. Ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτών των πραγμάτων. Ε, τώρα, ε, μιλήσαμε για το in προώθηση τη διαμεσολάβηση τη εκπαίδευση. Επίση, πιλωτικά προγράμματα και ευρωπαϊκά προγράμματα ε, διαμεσολάβηση, επίσης δέσμευση από τις εταιρείε ε, για τη διαμεσολάβηση και η ιδέα να βάλουμε εθνικούς πρεσβευτές, ε, δημόσια πρόσωπα, θα καλούσαν τους ανθρώπους, τους πολίτες να σκεφτούν τη δυνατότητα της διαμεσολάβηση. Προτάθηκε ακόμη και η Υπηρεσία ενολεκτικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν του Ινστιτούτου προ αυτή την κατεύθυνση. Οι εμπειρογνώμονε είπαν ότι θα λειτουργούσαν αυτά τα μέτρα, όμως θα ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών και σε οποιαδήποτε περίπτωση τα αριθμιστικά μέτρα είναι πολύ πιο σημαντικά. Και εδώ πηγαίνουμε στο εξή. Όταν συζητάμε την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, τότε ε, μπορεί να πάει κάποιος το άλογο στην πηγή, αλλά δεν μπορεί να το αναγκάσει να πιει. Δηλαδή, μπορείτε να οδηγήσετε τα μέρη ενώπιον του διαμεσολαβητή, αλλά δεν μπορείτε να τους αναγκάσετε τους διαδίκους ε, να βρουν μία λύση στα πλαίσια της διαμεσολάβησης. Ε, έτσι λοιπόν από τη σκοπιά της πολιτικής θεωρήθηκε άχρηστο. Δεν ε, νομίζω ότι οι πολιτικοί πρέπει να ανησυχούν για τον ε, εγώ χάνω το χρόνο μου για τη διαμεσολάβηση. Ένας πολιτικός θα έπρεπε να σκεφτεί ότι αν οδηγήσω 13 εκατομμύρια άλογα στην πηγή, στο ποτάμι, πόσα από αυτά τα άλογα θα πιούν και εκεί βάζω τη γραμμή, θα δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη των αλόγων που θα πιούν έναντι αυτών που δεν θα πιούν. Αν θέλεις να πιούν τα άλογα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα πιούν καλή ποιότητα ε, νερό και έχουμε και το θέμα της ποιότητας διαμεσολάβησης, αλλά τώρα δεν θα το συζητήσουμε. Τώρα, κάτι που ανέφερα προηγουμένως, έναντι μια επίθεσης ε, μπορεί κάποιος να σκεφτεί ε, την άσκηση μήνυσης, όμως ε, το ένστικτο του ανθρώπου είναι είτε να πολεμήσει είτε να φύγει. Και εγώ ξέρω ότι και στη φυσική ισχύει αυτό, δράση-αντίδραση. Αν ασκήσουμε μία δύναμη, έχουμε την απόθεση. Λέγεται και αμοιβαιότητα στην ανθρωπολογία και δράση-αντίδραση στη φυσική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και ένα νόμο ε, για να βάλουμε τη ζώνη ασφαλεία. Παίρνουμε το ξέρουμε ότι είναι καλό, αλλά έχουμε μία νομοθεσία που μα υποχρεώνει να φοράμε την ε, ζώνη όταν οδηγούμε και μα υποχρεώνει να φοράμε και κράνο. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλού νόμου που μα υποχρεώνουν να κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ως μέλη της κοινωνίας ότι ήταν καλό να το κάνουμε, αλλά αν δεν υπήρχε νομοθεσία δεν θα τα κάναμε. Αυτό είναι το νόημα εδώ. Επομένως, έχοντας ε, ε, δει το θέμα του παραδόξου, η τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης που υπάρχει και η αναποτελεσματικότητα των νομοθετικών μέτρων ή ε, των χαρακτηριστικών που υπάρχουν και Είδαμε τι είπαν και οι εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη σε σχέση με το τι είναι επιθυμητό και το τι χρειάζεται τώρα. Νομίζω ότι έρχονται δύο λύσει ε, κατά νου. Η πρώτη προσέγγιση θα ήταν να εισαγάγουμε ε, μία μετριασμένη υποχρεωτική διαμεσολάβηση στην οδηγία για τη διαμεσολάβηση και στα υπόλοιπα νομικά μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δύο επιλογέ. Η μία θα ήταν η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με opt-out, ε, δηλαδή να εγκαταλείψω τη διαδικασία με περιορισμένο κόστο ή χωρί καθόλου κόστο, αν δεν είμαι ικανοποιημένο, ή μία σύνοδο, δηλαδή να πρέπει να καθίσω με το δικηγόρο στη διαδικασία. Και από τα δύο ε, θα φαινόταν ότι η δυνατότητα του opt-out της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης είναι ανώτερη γιατί έχει μπορέσει να λύσει εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις στο τελικό μοντέλο σήμερα. Ενώ ε, στην ε, περίπτωση που έχουμε ένα διαφορετικό καθεστώς στην Τσεχία, στη Ρουμανία, στο Λουξεμβούργο, δεν ε, έχουν επιληθεί αρκετές περιπτώσεις και ζητείται κάτι ισχυρότερο από τους εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό η πρώτη λύση θα είναι η προτιμόμενη, όπως φαίνεται, χωρίς χωρίς να αναφερθούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Χωρί να αφήξουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που απαιτεί η λύση 1, η εναλλακτική που έχουν ε, τα κράτη θα ήταν ε, η αποκαλούμενη θεωρία της ε, ισορροπημένης σχέσης του αριθμού στόχου. Η θεωρία βασίζεται στο άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2008 που λέει ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας, δηλαδή να διευκολύνει την πρόσβαση σε εναλλακτική επίλυση διαφορών στη μεσολάβηση και διασφαλίζοντας Δηλαδή όχι να διασφαλίσει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών. Υπό τη θεωρία αυτή, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θέση να καθορίσει ποιος είναι ο δικός του στόχος και εδώ εννοούμε ένα ελάχιστο αριθμό υποθέσεων που θα λύνονται μέσω διαμεσολάβηση κάθε χρόνο έτσι ώστε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των υποθέσεων που πάνε στη διαμεσολάβηση και όσων πάνε στα δικαστήρια. Φυσικά, βάσει της αρχής της κάθε κράτος μέλος μπορεί να θέσει το δικό του στόχο και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα. Τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να εισαγάγουν την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να δώσουν απλώ οικονομικά κίνητρα. Αλλά αν δεν πετύχετε το στόχο αυτό εντό ενό έτου, δεν θα έχετε σεβαστεί την οδηγία. Είναι σαν τη συμφωνία του και όταν θέλουμε καλύτερο περιβάλλον πρέπει να πούμε πρέ, πόση ρήπανση πρέπει να περικόψουμε ή όπως συμβαίνει στην Ελίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Αν ε, δεν ξέρεις που πηγαίνεις, μπορείς να πας σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν ε, δεν ε, ξέρεις τι να περιμένεις, τότε έχουμε και ένα λόγια. Όμως, επειδή η διαμεσολάβηση πάντοτε θεωρούνται ένα αμερικανικό φαινόμενο, σήμερα όταν ε, λέμε ότι έχουμε μια δικαιοδοσία ε, ιδιαίτερα πολύπλοκη όπως ε, έχουμε στη Νέα Υόρκη το, δικαστήριο στο, το εμπορικό δικαστήριο στο Μανχάταν σκέφτεται να στην ίδια και από το Φεβρουάριο του 2014 και μετά κάθε νέα κάθε πέμπτη νέα υπόθεση θα αντιμετωπίζεται με τη διαμεσολάβηση. Έχουμε δηλαδή υποχρεωτική διαμεσολάβηση εδώ με το opt-out, γιατί έχει τη δυνατότητα ο διάδικος ε, να αποφευθεί στο δικαστή, να στραφεί στο δικαστή και να πει, ξέρω ότι είμαι, ε, είναι η σειρά μου, είναι η πέμπτη υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη υπόθεση αυτή για διαμεσολάβηση και κατά Όλα αυτά θα ήταν ακούσει. Έτσι λοιπόν, αν μιλήσουμε ορολογία Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να πούμε ότι η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει θέσει ένα στόχο στόχο 20% ε, για την εξισορροπημένη την σχέση θεωρία αυτή από την Ελλήνα Κάρθη ανακοινώθηκε πρώτα στην Επιτροπή αυτή τον Απρίλιο του 2012, δηλαδή δύο μήνες πριν από τους Αμερικανούς. Ευρωπαϊκή εφεύρεση λοιπόν. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα και φτάνω και προς το τέλος της παρουσίασης και ελπίζω ότι θα υπάρχει και χρόνος για ερωτήσεις. Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός. Χρειαζόμαστε μία μελέτη για να σκεφτούμε ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε διαμεσολάβηση είναι να κάνουμε τους πολίτες να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την επιλογή. Και να προσθέσω και μια άλλη οπτική, αν δείτε παγκοσμίω τι συμβαίνει, οι χώρε που έχουν κάποια υποχρεωτικά στοιχεία, δεν θα έλεγα περσέ υποχρεωτική διαμεσολάβηση, αλλά που έχουν κάποια στοιχεία, διατηρούν το σύστημα και το βελτιώνουν, δεν το εγκαταλείπουν. Ενώ οι χώρε που δεν έχουν κάτι τέτοιο σκέφτονται πώς θα το κάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι παγκόσμια είναι σαφή η τάση ω προ την πολιτική για τη διαμεσολάβηση. Και από τη Δανία, από το μύθο, για τον, παραμύθι για τον αυτογυμνό βασιλιά. Πάμε στο τελευταία διαφάνεια. Βλέπετε εδώ τη Στοκχόλμη, της 3 ε, Σεπτεμβρίου 1967, όταν η χώρα μετά από μια δημόσια διαδούλευση αποφάσισε ότι θα ε, αρχίσουν ε, να ε, ε, οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. Άλλαξαν το σύστημα λοιπόν οδήγηση. Ε, τι χρειάστηκε, εκπαίδευση και εμείς για τη διαμεσολάβηση είχαμε πάρα πολύ κατάρτιση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Απλώς χρειάζεται το θάρρος να πει κάποιος ότι από σήμερα και πέρα θα αλλάξουμε. Είναι δύσκολη η αλλαγή, αλλά είναι αυτό που χρειαζόμαστε και ελπίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα δώσει όθηση και υποστήριξη έτσι ώστε τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Αν και πρέπει να πω ότι κάποια πράγματα δεν είναι πολύ σαφή ως προς τις εξελίξεις για μένα. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να ασχοληθεί, να διευκρινίσει κάποια πράγματα σε σχέση με, την, με τα πραγματικά δεδομένα της διαμεσολάβησης. Ασφαλώς θα πρέπει κανείς να έχει συμφέρον να προχωρεί η διαμεσολάβηση όταν οι ε, διαδικασίες ενώπιον των δικαστήριων μπορεί να, κρατάν, να κρατούν ε, χρόνια. Άρα και οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον, όπω άλλωστε και οι δικηγόροι που μένουν ε, με εκκρεμότητε στους φακέλους τους για πολύ μακρύ διάστημα. Οι ασφαλιστικές εταιρείε, αλλά και τα δικαστήρια. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά τη προσφυγής στη διαμεσολάβηση. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να αξιολογήσουμε και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσφύγη στη διαμεσολάβηση. Οι συνάδελφοι έχουν ερωτήσει. Κυρία Τάιν. Ναι, ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Ως φιλελεύθερη, ομολογώ ότι προβληματίζομαι όταν ακούω προτάσεις για πράγματα που μπορεί να καταστούν υποχρεωτικά ή ιονή υποχρεωτικά. Και το ότι κάθε, κάθε πέντε υποθέσεις, τουλάχιστον με στατιστικές ε, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, όχι απαραίτητα υποχρεωτικά, σημαίνει ε, προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Δεν πολύ καταλαβαίνω αυτή την αναφορά. Πρέπει να αποφασίσουμε νομίζω ξεκάθαρα την κατεύθυνση που θα επιλέξουμε Φυσικά στο εμπορικό δίκαιο, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ τα πράγματα από το γερμανικό δίκαιο, έχουμε πολύ συχνή προσφυγή στα διαμεσολάβηση, το κατά πόσον ε, δείχνει επιτυχή εφαρμογή το σύστημα της διαμεσολάβησης στην Ιταλία, εκεί όπου είναι γνωστό πως ε, το δικαστικό σύστημα ε, σημαίνει και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και χρόνων καθυστερήσεις. Πάλι δεν με εκπλήσει. Από την άλλη, εμείς έχουμε προσπαθήσει στη Γερμανία με πολύ σοβαρές προσπάθειες και έχουμε καταφέρει να περικόψουμε τις ε, διαδικασίες μέχρι και μέσα σε δύο εβδομάδες έχουμε καταφέρει να έχουμε δικάσιμο και απόφαση μέσα στους δύο-τρεις μήνες. Άρα λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν βλέπω πολλά κίνητρα να καταφύγω εγώ στην διαμεσολάβηση, γιατί και αβέβαιο είναι το αποτέλεσμά της και βέβαια όταν πρόκειται ειδικά για πολλά χρήματα, άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα οικονομικό έρισμα. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τις περιπτώσεις στις οποίες ε, μπορεί να κοστίζει και πιο πολύ χρόνο η διαμεσολάβηση. Εγώ έχω παραδείγματι παραστεί σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης ε, ως δικηγόρος που αντί για το 1 τέταρτο που θα μου κόστιζε σε χρόνο η δικάσιμος, η εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, η παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, ε, χρειάστηκε να περάσω αρκετές ώρες για τη διαμεσολάβηση. Αυτό είναι ένα κίνητρο νομίζετε για τους δικηγόρους. Ή μήπως θα έπρεπε να αποφύγουμε τις υπερβολικές παραπομπές στη διαμεσολάβηση. ή μήπως πρέπει να κοιτάξουμε άλλα κίνητρα που ενδεχομένως οθούν του διαδίκου να καταφύγουν στη διαμεσολάβηση, όπως παραδείγμα το γεγονός ότι μπορούν να μιλούν από καρδίας ε, και δεν είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν του κανόνες κανόνε τη διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κάποια ε, ε, λύσεις οι οποίες θα καθιστούν πολύ πιο συμφέρουσα τη διαμεσολάβηση. Αλλιώς δεν θα δούμε κόσμο, ούτε δικαστές, ούτε διαδίκους, ούτε δικηγόρους να την προτιμούν. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, από πλευράς μου, για να συμπληρώσω μια ερώτηση, νομίζω ότι δεν είναι σε αντιδιαστολή η επιλογή μεταξύ δικαστηρίου και διαμεσολάβησης. Εγώ νομίζω ότι ε, πρέπει κανείς να κοιτάξει εάν είναι σοβαρή η προσέγγιση. Εμείς, ε, και θυμάμαι από τη δική μου την ε, υπηρεσία ως δικηγόρου, είχαμε πάντα σαν ε, κύριο μήνυμα, η κύρια ιδέα, το σύνθημα άμα κάνεις νωρίς την αγωγή έχει σχεδόν κερδίσει τη δίκη. αυτό ίσως είναι κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να δούμε και το πώς ε, δίνονται οι λύσεις στη διαμεσολάβηση και αν είναι σε αντιδιαστολή με αυτές τις δικαστικές διαδικασίες. Επίσης, ποιος μπορεί να είναι διαμεσολαβητής, ο ίδιος ο δικαστής. Και άρα είναι ίσως πιο οικονομικό ε, το γεγονός ότι ούτως, δηλαδή είναι οικονομικά πιο συμφέρον το γεγονός ότι ούτως ή πρέπει να διαβάσει το φάκελο της υπόθεσης και να λάβει μια απόφαση, όπως το έκανα και στην έδρα. Ή αλλιώς μπορεί να υπάρχουν άλλες δομές στα κράτη-μέλη. Επί παραδείγματι υπάρχει ένα σύστημα παροχής ε, διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στη Γερμανία το οποίο λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλές ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά όπως τις άκουσα. Και καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είμαι υπέρ της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης αυτής καθεύτης. Όταν βλέπω προσφυγή σε μένα με, στόχο, με εθελοντική αυτοδέσμευση των μερών, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ πιο ένθερμος. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχει αποτύχει κάθε σύστημα, ακόμα και το οικονομικό κίνητρο στις χώρες που το χρησιμοποίησαν και δεν έχει λειτουργήσει αρκετά ελκυστικά το σύστημα. Άρα λοιπόν, ειδικά για χώρες που δεν έχουν μεγάλα πλούτη, δεν ε, τους περισσεύουν τα λεφτά, δεν είναι λύση το οικονομικό κίνητρο. Σαν απάντηση μπορώ να σας δώσω ότι το αμερικανικό σύστημα μπορεί να είναι κάπως αυτόματο, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι η πέμπτη στη σειρά υπόθεση που θα, θα, θα φτάσει στα δικαστήρια είναι ε, πρόσφοροι για διαμεσολάβηση. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα. Φερρυπίν στην Ιταλία, πρέπει να δούμε, ε, υπάρχουν ε, αποτελέσματα, έχουμε μια κατηγορία διαφορών που είναι πιο πρόσφορες για τη διαμεσολάβηση. Να κοιτάξουμε για τις κληρονομικές διαδοχές, για ενδεχομένες αγωγές, για ιατρικό σφάλμα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα καταγράψουμε και να δούμε πώς αποδίδει το σύστημα. Όταν βέβαια το σύστημα της προσφυγής στη δικαιοσύνη, την παραδοσιακή, ε, δεν λειτουργεί, κρατάει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή, ίσως πρέπει κανείς να προχωρήσει τη μεσολάβηση. Από την άλλη, αν το νομικό μου σύστημα είναι πάντα υπέρ του οφειλέτη, εκείνο δηλαδή που αρνείται τελικά να πληρώσει ή δεν ε, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, ποιος έχει συμφέρον να πάει στη μεσολάβηση. Για δε την διάρκεια των διαδικασιών σας διαβεβαιώ ότι και οι δικηγόροι και οι δικαστές δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ε, για τις παρατηρήσεις ότι η διαμεσολάβηση, ε, έστω και αν εγώ επικεντρώθηκα στο χρόνο σαν παράγοντα που την καθιστά ενδιαφέροντα, δεν έχει μόνο αυτό το πλεονέκτημα να προσφέρει. Γιατί δεν μπορεί κανείς να φρενάρει το άλογο όποτε ε, πατήσει το σπιρούνι η τραβήξη χαλινάρι. Ωστόσο υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να προσφέρει η διαμεσολάβηση, την, ε, την πιο συμβιλιωτική διάθεση και όλα αυτά που μπορούμε να τα ε, αξιοποιήσουμε. Για την ε, δική σας παρατήρηση κύριε Πρόεδρε, η διαφορά μεταξύ διαμεσολάβησης και διαιτησίας ίσως είναι απαραίτητο να κριθεί με βάση το κατά πόσον θα είναι δεσμευτική η συνέχεια της διαδικασίας, η διαφορά δηλαδή με την διαιτησία. Δεν αναιρεί την, δια, την διατησία, η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα όλο μαζί της. Αυτό που είπατε για τους ε, δικαστές που αναλαμβάνουν και ως διαμεσολαβητές καθήκοντα έχει αξιοποιηθεί κυρίως στις χώρες ε, της Βόρειας Ευρώπης. Έχει ένα πλεονέκτημα ασφαλώς γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μελετήσει το φάκελο ο δικαστής. Από την άλλη διατρέχουμε και τον κίνδυνο να ε, προκύπτει σε περίπτωση που μετά επιληφθεί τις ίδιες υπόθεση να υπάρχει μια ε, προεξόφληση του, της ετοιμιγορίας του η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ε, και έτσι μια λύση θα μπορούσε ο δικαστής όταν έχει διαμεσολευήσει σε μια υπόθεση να μην κάθεται στην έδρα για την ίδια υπόθεση Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις δηλαδή. Τα συστήματα μπορούν να προχωρήσουν και πιο γρήγορα. Σίγουρα μαζί. Ευχαριστώ πολύ. άλλε ερωτήσει, λέει ο πρόεδρο. Όχι, σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. περίπλοκα νομοθετήματα αυτά που θα χρειαστεί να υιοθετηθούν για την ε, διαμεσολάβηση. Εσφαλώ δεν θα προλάβουμε στην τρέχουσα θητεία, αλλά ελπίζουμε στην επόμενη να τα δούμε. Βλέπω ότι δεν έχουμε ακόμη, για να περάσω το επόμενο θέμα, δεν έχουμε ακόμη απαρτία. Προχωρώ. Ανακοινώσει του Προέδρου, στο 2 της σημερινής διάταξης. Ξεκινάμε 3.30 αύριο και όχι 3 τη συνεδρίασή μας. Αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να, δηλώσω, να ανακοινώσω.